κατόπιν επαλήθευσης των γεγονότων και περνάω πια στην ψηφοφορία. Πρώτον, η διάσκεψη των Προέδρων έχει προτείνει στο Σώμα την παράταση της εντολής της ε, ε, Επιτροπής για την ε, ε, διερεύνηση φορολογικών πρακτικών και άλλων της τάξης 2 να έως τον Αύγουστο του 2016 υπάρχουν αντιρρήσεις όχι άρα θεωρούμε ότι εγκρίνεται και προχωρώ στην ψηφοφορία στα ρωμανικά μάλιστα Πρώτον, πρώτη έκθεση, ελευθερία της έκφρασης στο Καζακστάν το ψήφισμα. Τροπολογία 5 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 12, παράγραφος 12, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, υπέρ, κάτω. Αποχές, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία δεύτερη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τρία. Ονομαστικά. Αρχίζει ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στο ψήφισμα το σχετικό με την Αίγυπτο και ιδίως την υπόθεση Τζούλιο Ρετζένη. Σημείο, ε, 3 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. κρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία τρίτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη.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 Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απερίφθη. Το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Πέρασε Εγκρίνεται. Λογοκρατική Δημοκρατία του Κόγκο. 7 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε όμως. Αρχίζει η Πέρας. Και απερίφθη. 8 υπέρ. Ναι. Κατά. Και αποχές. Νομίζω ότι οι πλειοψηφίες είναι οι ίδιες. Απερίφθη δηλαδή. Δεύτερη τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Άποχες. Επαληθεύουμε. Και η ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10 στο αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 3 υπέρ κατά άποχες απεριφθεί τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές και απερίφθη τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και συνεχίζουμε Έφεστε σαρνές ε, για τη θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τινησία. Μία ψηφοφορία, ονομαστική όμω. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, έκθεση Φρανσουάς Γκροστέτ, κτηνιατρικά φάρμακα. Έχουμε πολλές τροπολογίες. Από την Επιτροπή που τις ψηφίζουμε από κοινού υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνονται αυτές οι τροπολογίες. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Καλώς, άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 49. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 74, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 291 ονομαστικά Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. απορρίπτεται. Τροπολογία 77, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 297D, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 99, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 100, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.92-3.15 ταυτόσημες με ονομαστική... Α, καταπίπτουν. Πάμε στην 3.16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 3.16. Τροπολογία 111 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 112, ψήφι περ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Τροπολογία 113, πρώτο τμήμα, ψήφι περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 293 ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 116 ψήφι ΠΕΡ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 298 D. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 κατά τμήματα. Όχι, θέλετε να ελέγξουμε την προηγούμενη τροπολογία. 298 διάρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. με ακούλπα. Τροπολογία 117 πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 127. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. 127 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 131. Ονομαστικά ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Έχετε ένα πρόβλημα μήπως? Εκτός μικροφώνου. Υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω της ε, διερμηνίας. Εντάξει, θα προσπαθήσω να μην μιλάω τόσο γρήγορα. Να κρατάω κάποια απόσταση από μια εκφώνηση ψήφου Δεν είναι παρελκυστική τακτική για να καθυστερήσουμε. Όλοι έχουμε αεροπλάνα ή τρένα να προλάβουμε. Και αυτοί και οι άλλοι συνάδελφοι. 131. Ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 299 τροπολογία ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 300. Ονομαστική άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην ονομαστική ψηφοφορία. Και εγκρίνεται ονομαστικά τώρα πέρας απορρίπτεται δεν βλέπω τα φώτα ε, στη, στα μηχανήματα γι' αυτό και συνεχίζω 318. 319. Ε, ονομαστική άρχεται. Votul este închis. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. 312 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 137 καταπίπτει. 138. Κατά. Εγκρίνεται. Η 320 καταπίπτει. 300, 321 συνομένα μαστικά. Και πέρας. Απερίφθη. 322 ονομαστικά αρχής ψηφοφορία πέρας απερίφθη 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 και πάλι υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται 144 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απερίφθη 144 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ένωση της ψηφοφορίας για το 144 θα κάνουμε ηλεκτρονική υπαλλήθευση. Πέρας. Και εγκρίνεται. Έκανα λάθος εγώ, λέει ο πρόεδρος. Σούτα Πατρουζέτσι. 150. 150. Cine este... 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151. Ονομαστική. Ψηφίσμα. Πέρας. Εγκρίνεται. 152. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Ας κάνουμε επαλήθευση για την 152. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 186. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εγκρίνεται. Θεωρώ ότι έχει εγκριθεί. Και πάμε επομένως στο 202. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 302 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται 213 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα αποχές θα γίνει η επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα του 213 ψηφίζουμε πέρασε 317 ονομαστική ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 226 ονομαστική ψηφίζουμε. Πέρας. και εγκρίνεται. 2.27 ονομαστική ψηφίζουμε. Πέρασε. και ονομαστική ψηφίζουμε. Votul este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 και 108 καταβίβουν και πάμε στο 234 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα και ηλεκτρονικά θα επαληθεύσουμε για το 234 πέρας εγκρίνεται 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εγκρίνεται. 303 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για το 303 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 48. Καταπίπτει. 250. Υπέρ. Τις 250 παρακαλώ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 304 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 253 καταπέφτει. Πάμε στη 254 με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 262 ψηφίπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.73 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.78 με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 305. Με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 283 ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 306 καταπίπτει. 307 με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 308 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 309 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 310 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 290 ψηφίπερ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 6 ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία τώρα 313 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.14 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 καταπίπτει η 296 ρεπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε η κυρία Γκροστέτε ζητεί το λόγο παρακαλώ έχετε το λόγο κυρία Γκροστέτε θα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα κύριε Γκροστέτ έχετε παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Προτείνω αναπομπή, ε, μάλλον ε, αναβολή ε, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού να αναβάλουμε την ψήφιση ε, του νομοθετικού ψηφίσματος για να προχωρήσουμε αμέσως σε διαπραγματεύσεις βάση της εντολής ε, που μόλις λάβαμε. Ο Πρόεδρος. Θα πρέπει να ψηφίσουμε την πρόταση αυτή ε, με ονομαστική κλίση ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα. Is closed. Εγκρίθηκε. Ne ducem mai departe la Ευχαριστώ. Ακολουθεί τώρα η έκθεση του κυρίου Τανασέσκου. Και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Όχι. Δεν επιθυμεί ο εισηγητής να λάβει το λόγο. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Ε, λάθος χαρτιά έχω. Ε, έχουμε unblock τις τροπολογίες της ε, Αρμόδιας Επιτροπής 1 ε, με 35. Ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Θανασέσκου. Ευχαριστώ. Προτείνω να υπερψηφίσετε την πρόταση βάσει των κανόνων για τις ε, διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις ε, για την εντολή. Παρακαλώ ψηφίζουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τώρα, Ε, το επόμενο θέμα για μια ε, οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα. Πρώτο απολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το τμήμα 2 υπέρ. Το δεύτερο καταπίπτει. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το πρωτότυπο τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 παράγραφος πρωτότυπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 26 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές Εξακρίβωση. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το τμήμα 2 της παραγράφου 26 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παραγράφος 29. Τμήμα 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραγράφος 36. Τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τη λογική σκέψη β. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. λογική σκέψη C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. λογική σκέψη D τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το επόμενο σημείο είναι η κατάσταση στην Ερυθρέα. Ε, έξι, το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία υπέρ. Ε, άρχιτη ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τμήμα 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16 τμήμα 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η έκθεση για την ε, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ε, τροπολογία είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, παράγραφος είναι υπέρ. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, για την 7 θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 32, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Α, θα γίνει μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Όχι, ζητά συγγνώμη πρόεδρος. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 με ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 45. Το πρωτότυπο πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Τμή πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τμήμα 2 Καταπίπτει. Ε, παράγραφος 48. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρι... Εγκρίνεται. 17 αντί με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται και πέρας. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ κατά αποχές ελεγχός άρχεται για την ε, τροπολογία 8 πέρας εγκρίνεται ε, ε, τροπολογία είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η ε, σκέψη σύμφωνα είναι υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, η 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τετελογική σκέψη G. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Ήταν ε, ε, προφανές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ακούσατε τη μετάφραση από τα ρουμανικά, κύριε Μαριά. Πέραση ψηφοφορίας. Εντάξει, υπήρχε μία μικρή διαφορά που δεν φαίνεται από εκεί πάνω. Τώρα πάμε στην έκθεση για το Μαυροβούνιο. Αμενταμέντο 6. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπάρχει κράτος. τροπολογία τροπολογία 7 και 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ε, για τις 4 και 7 άρχεται πέρας εγκρίνεται Συγγνώμη, έκανα λάθος, έχω να καθαρίσω τα γυαλιά μου, δεν βλέπω καλά. 9. απολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 33 ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας Εγκρίθηκε. Τροπολογία είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κύριε Κόβατσεφ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα από πλευρά του ΕΛΚ να υποβάλω μια προφορική τροπολογία, τροπολογία 3, πρώτο τμήμα, μετά την πρώτη πρόταση. Ε, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ε, ε, εξωτερικές πιέσεις σε σχέση με την συμμετοχή του Μαυροβουνίου στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Πρόεδρος, υπάρχουν αστάσεις? Όχι. Έχουμε 40 συναδέλφους που αντιτάσσονται στην προφορική τροπολογία. Συγγνώμη. Θα ε, ψηφίσουμε για το πρώτο τμήμα όπως είχε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. τμήμα 2 της ε, τροπολογίας 3. Θέλετε αυτό. Ωραία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται δύο Η δύο καταπίπτει. Το πρωτότυπο κείμενο. Πρώτο Όχι, για το σύνολο του ψηφίσματος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. μια συμβαστική τροπολογία από πλευρά του κ. Ε, πολύ αργοπορημένα την έλαβα και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν ενστάσεις. Όχι. Θα ψηφίσουμε για τροπολογία 1 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Μια ανακοίνωση ζήτησε χωριστή ψηφοφορία για την ε, παράγραφο 50. Όμως αποσύρθηκε η παράγραφος και τόσο σέλος δεν θα ψηφίσουμε. Γι' αυτό περνάμε στην παράγραφο 64 με νομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 65 με νομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 66. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Για το σύνολο του ψηφίσματος, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ. Θα παραμείνω εγώ για τις υπεξηγήσεις ψήφου. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να αποχωρήσουν ε, γρήγορα και αθόρυβα από το ημικύκλιο, παρακαλώ. Colegi, putem trece la explicațiile de vot. Ακολουθούν επεξηγήσεις ψήφου τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζεται η συζήτηση. Παρακαλώ, έχουμε τις επεξηγήσεις ψήφου τώρα.